Mes chers collègues, je vous remercie pour votre présence pour notre réunion de commission. Καλώς ορίσατε ε, κυρίες και κύριοι στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας σήμερα το βράδυ στο Στρασβούργο. Πριν ε, έλθω στο θέμα που θα μας απασχολήσει, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των ε, συναδέλφων που συμμετείχαν στην Εβδομάδα των Περιφερειών, μια εβδομάδα πολύ πλούσια σε εκδηλώσεις και γεγονότα. Ήταν μια σημαντική στιγμή γιατί μπορέσαμε να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί και να ε, επιχειρηματολογήσουμε υπέρ της συνοχής σε ένα μέλλον το οποίο είναι απολύτως ε, σημαντικό και κρίσιμο για τη δική μας πολιτική. Συνεδριάζουμε λοιπόν σήμερα για την ψηφοφορία, για την τροποποίηση του κανονισμού που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Αλληλεγγύης, προκειμένου πρώτον και σωστό θυμίζω να προσθεθεί το Brexit στις ε, συνθήκες που τεκμηριώνουν την ανάγκη εκταμίευσης ε, κονδυλίων από το Ταμείο, διότι το Ταμείο αυτή τη στιγμή καλύπτει μόνο τις φυσικές καταστροφές και δεύτερον να ψηφίσουμε να αυξηθούν από 10 σε 25% οι προκαταβολές και για τις φυσικές ε, καταστροφές και για το Brexit. Η Επιτροπή Προϋπολογισμού εξέτασε την πρόταση αυτή και έχει εκδώσει μια γνωμοδότηση με τη μορφή επιστολής η οποία διάκειται θετικός. Ε, ως προς την πρόταση αυτή. Στην Επιτροπή Ρέτζι το συζητήσαμε στις 2 Οκτωβρίου και η πρόταση υιοθέτηση της απλουστεμένης διαδικασίας δεν εγκρίθηκε. Την επομένη οι συντονιστές επομένως αποφάσισαν να μου αναθέσουν αυτό το φάκελο βάσει της τακτής διαδικασίας. Όμως λόγω του επίγοντος χαρακτήρα ακολουθήσαμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο ήταν όσο το να δω πιο περιορισμένο. 87 τροπολογίες έχουν, έχουν υποβληθεί και την περασμένη εβδομάδα έχουμε συμφωνήσει πάνω σε τέσσερις συμβεβαστικές τροπολογίες που καλύπτουν τα πιο σημαντικά σημεία της πρότασης. πρότασης. Η έκτακτη συνεδρίαση λοιπόν σήμερα το βράδυ έχει ως ε, στόχο να ε, ψηφίσουμε τις τροπολογίες και το φάκελο αυτό, γιατί ο φάκελος αυτός θα ε, ε, είναι στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειάς μας. Προτείνω λοιπόν να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία πριν μετά την ψηφοφορία να συζητήσουμε τα διαδικαστικά θέματα στην Ολομέλεια και για τη συνέχεια που μπορούμε να επιφυλάξουμε στο φάκελο αυτό. Να ψηφίσουμε δηλαδή πρώτα και να συζητήσουμε τα διαδικαστικά στη συνέχεια, γιατί ήθελα να σας θυμίσω το εξή. Ο κανονισμός που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αφορά σε μια υπόθεση εργασίας, στην υπόθεση του Brexit χωρίς συμφωνία, στο no deal, στην περίπτωση στην οποία δεν θα υπάρχει συμφωνία. Και ε, Κανεί δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή εάν στι 31 Οκτωβρίου θα έχουμε deal ή θα έχουμε no deal. Μπορεί κανείς να κάνει τις υποθέσεις του, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος. Άρα η ευθύνη μας ως νομοθέτες, όπως σας έχω ήδη αναφέρει, είναι να ε, προετοιμαστούμε για παν ενδεχόμενο. Εξού και είναι ανάγκη να γίνει αυτή η ψηφοφορία. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε ευθύ αμέσω και να ε, συνεχίσουμε στη συνέχεια. Έχετε τις κάρτες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, τις έχετε βάλει στο μηχάνημα. Να κάνουμε μια επαλήθευση μπορούμε, από ό,τι βλέπω όλα καλά, άρα μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία για την πρόταση της απόρριψης του κανονισμού ο οποίος καλύπτει μια σειρά, ε, πρόταση η οποία καλύπτει μια σειρά τροπολογιών που βρίσκονται στον κατάλογο ψηφοφορίας που έχετε μπροστά σας. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία. Τώρα λοιπόν θα περάσουμε στο 3 Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, η τροπολογία, οι τροπολογίες απορρίπτονται. Και τώρα περνούμε στην ψήφιση του συνόλου των τροπολογιών, δηλαδή των τροπολογιών από την 37 ως και την 33. 33 με 37 τις ψηφίζουμε από κοινού λέει ο πρόεδρος. Ναι. Συγγνώμη. Συμβιβαστική 1. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Ψηφίζουμε αυτήν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Εγκρίνεται η Συμβιβαστική τροπολογία 1. Περνούμε στη Συμβιβαστική τροπολογία 2 ποιο είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται η συμβιβαστική τροπολογία. Περνούμε στην τροπολογία 55 συναδέλφου Βάνα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε τη συμβιβαστική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Περνούμε τώρα στη ψηφοφορία της τροπολογίας 61. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να το θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται. Καλώς. Θέλετε να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 64. Παρακαλώ. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 65. 66, συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71 και 76 μαζί τις ψηφίζουμε. 70 και 71 και 76 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Α, καταπέπτει, καταπίπτει, συγγνώμη. Άρα πάμε στην 74. Ποιος είναι υπέρ? 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Την 80 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη ψηλιοψηφία. Τροπολογία 81. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, καταπίπτει. Άρα για 25, άρα για την τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται η έκθεση αυτή με 33 ψήφους υπέρ, καμία κατά, τέσσερις αποχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να σας δώσω κάποιες ενδείξεις, κάποιες ε, οδηγίες για τη διαδικασία στην Ολομέλεια. Καταρχάς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας γνωστοποίησε το ότι προς το παρεόν μεταθέτει χρονικά την εξέταση αυτού του φακέλου μέχρι <laughs> ότου διευκρινιστούν οι συνθήκες του Brexit. Όμως, άπαξ και γίνουν πιο σαφείς οι συνθήκες αυτές, αυτή η πρόταση θα μπορούσε να αποκτήσει έναν κατεπήγοντα χαρακτήρα. Και όπως σας το έλεγα, ήταν δική μας ευθύνη να οπλιστούμε ε, για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε παν ενδεχόμενο. Προβλέψαμε λοιπόν την εξέταση της έκθεσης και την ψήφιση της στην Ολομέλεια την Πέμπτη, εάν συμφωνείτε. Λοιπόν, θα ζητήσω την εφαρμογή του άρθρου 59 τέταρτη παραγράφου, τέταρτου εδαφίου του κανονισμού, ο οποίος λέει τα εξή και παραθέτω. Εάν το σύνολο του σχεδίου νομοθετικής πράξης εγκρίνεται, ο πρόεδρος αναγγέλει ότι κλείνει η πρώτη αγνάγνωση, εκτός και αν κατόπιν πρότασης του Προέδρου ή του εισηγητή της αρμόδιας κοινοβουλευτική Επιτροπής, αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραπέμψει το θέμα στην αρμόδια Επιτροπή με σκοπό να υπάρξουν διαθεσμικές και διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει των άρθρων 60 και 74. Πράγμα το οποίο προτίθεμαι να πράξω. Διότι η διαδικασία αυτή συνδυάζει διάφορα πλεονεκτήματα. Η Ολομέλεια υιοθετεί μία θέση με επίσημη ψηφοφορία Στη συνέχεια διαπραγματεύσεις γίνονται εφικτές και δυνατές τους τέσσερις μήνες που θα ακολουθήσουν, άρα δεν είναι απαραίτητο να εγκριθεί εντολή συγκεκριμένη κατά τη διάρκεια αυτής της έκτακτης συνεδρίασης. Και μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε να προχωρούμε εάν το απαιτήσει αυτό η, η εκάστοτε κατάσταση. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την ανακοίνωση της εντολής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Νοεμβρίου πριν ξεκινήσουμε τις ε, ενδυνάμει διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι η λύση αυτή μας ταιριάζει ανεξαρτήτως της ε, λύσης που θα θετηθεί για το Brexit τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Άρα, θα ζητήσω το λόγο μετά την ψηφοφορία για να πω ότι ζητώ να ε, παραπέμψουμε το φάκελο ε, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει με το Brexit. Δική μου πεποίθηση. Δεν βάζω στοίχημα βέβαια, αλλά δική μου πεποίθηση είναι ότι υπάρχει πολύ ασθενής πιθανότητα να υπάρξει Brexit χωρίς καμία συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει βάλει ένα επιτάπητος μία πρόταση για deal. Περιμένουμε να μάθουμε τη θέση των Βρετανών. Πιστεύω όμως ότι στα διάφορα σενάρια που διαμορφώνονται, το σενάριο του Brexit χωρίς καμία συμφωνία είναι το πιο ισχνό. Θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτή τη δουλειά και πιστεύω ότι οι τροπολογίες που έχουμε υποβάλει μας επιτρέπουν να διατρανώσουμε την ε, προσήλωσή μας στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Είδατε ότι μας ε, ότι έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στις φυσικές καταστροφές που έχουν πλήξει την Ισπανία και την Πορτογαλία. Ήμουν στη συνεδρίαση στη Σικελία στο Παλέρμο και ε, συναντήθηκα με τον πρόεδρο της περιοχής των Αζόρων Νήσων, με τον κυκλώνα, τον Λεωνάρντο, ο οποίος έπληξε την περιοχή και οδήγησε σε καταστροφές, προκάλεσε καταστροφές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν καταστραφεί όλες οι λιμενικές υποδομές της αζόρε μεταξύ άλλων και οι τροπολογίες που ψηφίσαμε επιτρέπουν μεταξύ άλλων να ε, υπάρξει η αναγκαία ισορροπία και η αναγκαία ενίσχυση του Ταμείου αλληλεγγύης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι φυσικές καταστροφές μάλλον και δυστυχώς θα πολλαπλασιάζονται προϊόντος του χρόνου. Όπως το γνωρίζετε, ε, σήμερα το, σήμερα το βράδυ συνεδριάζει η διάσκεψη των Προέδρων για να συζητήσει το Brexit. Ενδεχομένως μας καλέσουν στην Ολομέλεια πριν από τα τέλη Οκτωβρίου. Αύριο το απόγευμα υπάρχει μια συνεδρίαση μεταξύ των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και θα σας στηρώ ενήμερους και ενήμερες για την εξέλιξη της κατάστασης. Και αν η κατάσταση εξελιχθεί ε, δραστικά ε, μέχρι την Πέμπτη, τότε θα πρέπει να υποβάλουμε και εμείς σχετικό αίτημα. Σε κάθε περίπτωση ε, προς το παρόν προχωρούμε φυσιολογικά, κανονικά, πηγαίνουμε στην Ολομέλεια και έχουμε το φάκελο στην Επιτροπή μας και στη συνέχεια θα δούμε ποια συνέχεια αρμόζει καλύτερα να δώσουμε αναλόγως με το πώς θα έχει εξελιχθεί και η κατάσταση. Αυτά λοιπόν είχα να πω. Αν θέλουν οι σκιώδεις εισηγητές να πάρουν το λόγο, τώρα είναι η στιγμή. Για το ΕΛΚ, για τους σοσιαλιστές, για τους, ε, σε άλλες πολιτικές ομάδες, θέλει κάποιος σκιώδης εισηγητής ε, το λόγο. Από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, από τους πράσινους, από την ΚΟΕ. Ναι, κάτι μικροφωνίζει πράγματι και μας δυσαρεστεί αυτό. Είναι πολύ δυστυχές και δυσάρεστο. Est-ce que les services techniques peuvent régler ce problème? Δεν ξέρω, οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν κάτι να κάνουν, να μην μικροφωνίζει τόσο. Très bien. Bien. Bon, euh, autre chose. Puisque nous Καλώς, κάτι άλλο. Αφού είμαστε εδώ, ας συζητήσουμε λίγο την κατάσταση. Είδατε ότι συνεδρίασε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εγώ ήμουν στο Παλέρμο με τον συνάδελφο τον Γιάνν Όλμπριχτ και τον συνάδελφο από την Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών, την κυρία δηλαδή Μαργαρίτα Μάρκες, και από το Παλέρμο μπορέσαμε να αντιδράσουμε για τις προτάσεις που είναι ε, ε, αυτή τη στιγμή επιτάπητος και προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι προτάσεις μειώσεων περικοπών σημαντικών για το προϋπολογισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής και για το προϋπολογισμό της ε, πολιτικής συνοχής. Και από το Παλέρμο, με τους συναδέλφους από την Επιτροπή ε, Προϋπολογισμού, Υιοθετήσαμε ένα δημόσιο λόγο συγκεκριμένο, ο οποίος θεωρώ ότι είναι η θέση της Επιτροπής μας. Ότι δηλαδή αρνούμαστε αυτές τις περικοπές, αυτές τις μειώσεις. Θα σας πω λοιπόν ότι ήδη από αύριο στη συνεδρίαση των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Θα προτείνω στο σύνολο των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών να υιοθετήσουν τον ίδιο δημόσιο λόγο απευθυνόμενοι προς το Συμβούλιο. Δηλαδή όχι μόνο η Επιτροπή για τον Προϋπολογισμό και όχι μόνο η Επιτροπή Ρέτζι, οι δύο δικές μας, αλλά οι όλοι οι πρόεδροι όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Και αυτό θα προτείνω και στον πρόεδρο Ταγιάννη, γιατί πιστεύω ότι η διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών πρέπει να είναι ένα όργανο που να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις και ε, πολιτικές θέσεις. Και πρέπει λοιπόν να εθετήσουμε θέσεις σε σχέση με το ε, CFP. Σας ζητώ λοιπόν όλοι εσείς να αντιδράτε δημόσιο σε κάθε ευκαιρία και να υπερασπίζεστε την ανάγκη Προστασία του προπολογισμού. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στι διαπραγματεύσει για τους διάφορους κανονισμούς και αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε και να το καταφέρουμε εάν δεν έχουμε και αντίστοιχο προπολογισμό. Χωρίς αντίστοιχο προπολογισμό, θα δυσκολευτούμε ιδιαίτερω να εφαρμόσουμε μια καλή πολιτική, ειδικά για τα χρόνια που ε, έρχονται. Και όπως το είπα και στον πρόεδρο των περιφερειών, πρέπει κανείς να θετεί δημόσιο λόγο, πρέπει να είναι ενεργός στο Twitter, πρέπει να απευθύνεται στους διαφόρους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση. Τώρα, ως προς την κοινή γεωργική πολιτική και την πολιτική συνοχής, να σας πω ότι ε, δεν είναι η ίδια οργάνωση και ούτε οι δικαιούχοι. Η επικοινωνία είναι πολύ δυσάρεστο, το ξέρω αυτό με τον ήχο. Θα ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση κάπου εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και εμείς. Είναι πολύ δυστυχές και το δυσάρεστο στρέφουμε προς τον τεχνικό για να του το πω, λέει ο Πρόεδρος. Είναι πολύ κρίμα. Καλώς, ευχαριστώ όλους και όλες.